που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο στη Γεωργία. Η ΕΦΣΑ, τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία ασχολούνται με τις δραστικές αυτές ουσίες που δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν οι αγρότες τα παράσιτα κατά πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτό ε, θα σήμαινε ότι έχουμε και μία καλύτερη αποτίμηση τοξικολογίας αυτών των προϊόντων. Πιστεύω ότι η βιώσιμη αυτή χρήση παρασιτοκτόνων θα πρέπει να ενταχθεί στην ΚΑΠ. Θα είδατε ότι οι διατάξεις αυτές εντάσσονται στην πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα να υποστηρίξετε αυτή την έκθεση. Μετά από πέντε χρόνια από την εφαρμογή των πρώτων σχεδίων, εθνικών σχεδίων δράσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Εμείς θα υποβάλουμε μια δεύτερη έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας βιώσιμης χρήσης αργότερα φέτος για να αναθεωρηθούν και τα εθνικά προγράμματα δράσης και να οριστούν οι αδυναμίες. Επίσης θα δούμε ποια είναι η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Θεωρούμε ότι η οδηγία για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί ε, αναπόσπαστο στοιχείο της ΚΑΠ. Δύο εβδομάδες πριν συντάξαμε ένα έγγραφο για την βιώσιμη χρήση αυτών των προϊόντων μέχρι το 2020. Αυτό αφορά και τη διανομή και την κατανάλωση και αυτά δηλαδή τα δίκτυα. Και πιστεύουμε ότι η βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων θα βοηθήσει σε αυτό. Θα έχουμε και συστάσεις με βάση την έκθεσή σας. Η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε να εφαρμοστεί πλήρως αυτή η οδηγία και θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για την επίτευξη του στόχου αυτού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Οι πολιτικές ομάδες τώρα, με μια καθυστέρηση, άρα μπλε κάρτες δεν ε, γίνονται δεκτές στη φάση αυτή. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κ. Φλόρεντς, 1,5 λεπτά. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δεν μπορώ παρά να στηρίξω αυτά που είπατε. Μ' αρέσει γενικά η κατεύθυνση αυτής της έκθεσης. Το σημαντικό είναι το θέμα της περαιτέρω και συνεχούς κατάρτισης των γεωργών που χρησιμοποιούν αυτούς τους ε, ψεκαστικούς μηχανισμούς. Ε, εγώ έκανα με τέτοια κατάρτιση το Δεκέμβριο, παρά το ότι έχω και τρει άλλου εργαζόμενου που μπορούν να κάνουν αυτόν τον ε, ψεκασμό. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί και περισσότερο η αντίστοιχη τεχνολογία. Ε, συμφωνώ, μάλιστα ως ε, ενεργός γεωργός. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, έγραψε πολλά πράγματα από καρδίας και συζητούμε για το πώς θα υπάρξει βιώσιμη γεωργία. Δεν συζητάμε για την μόλυνση, για παράδειγμα, των υδροφόρων οριζόντων. Αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι όσο και εσείς και εγώ βεβαίως θέλουμε να έχουμε φθηνό κρέας, τότε να μην ε, ε, ε, αρνείστε να καταλάβετε κάτι. Κοιτάξτε, ε, ο πατέρας μου ε, είχε 28 ε, χείρους. Εγώ έχω 800 και η επόμενη γενιά θα έχει 3.000. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για βιώσιμη γεωργία αν έχουμε τέτοιες εκμεταλλεύσεις. Βεβαίως, κύριε Επίτροπε, απαγορεύουμε τα νεονικοτινοειδή. Αλλά εάν υπάρχουν 20 εξαιρέσεις, τότε στην ουσία υπονομεύουμε τα κράτη που εφαρμόζουν αυτή την απαγόρευση και ενθαρρύνουμε αυτούς που δεν την εφαρμόζουν. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, Πάβελ Τότς. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκιούτελαντ ε, ε, συνέταξε μια θαυμάσια έκθεση. <clears throat> Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το κάνουν. Η ολοκληρωμένη χρήση των, ε, αντιμετώπιση συγγνώμη, των ε, παρασίτων ε, είναι κάτι που είναι καθήκον των κρατών μελών του 2014 αλλά δεν το κάνουν και μας λένε παραμύθια. Δεν πρέπει να πάρουμε τα εργαλεία από τα χέρια των γεωργών. Πρέπει να τους δώσουμε αυτά που είναι κατάλληλα για την υγεία μας και για το περιβάλλον. Τα χημικά παρασυνοκτόνα και η χρήση αντιβιωτικών αυτό θα πρέπει να είναι μόνο ίστατη καταφυγή για τους γεωργούς και όχι το πρώτο μέσο το οποίο χρησιμοποιούν οι γεωργοί μας. Γι' αυτό λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχθηκε την πρόταση του Κοινοβουλίου να περάσουμε ταχύτερα στα πιο ακίνδυνα παραστοκτόνα. Θα χρειαστεί να περιμένουμε την επόμενη περίοδο φαίνεται. Πολύ συχνά μιλάμε για ασφάλεια, αλλά στην ουσία βάζουμε μια ορολογιακή βόμβα στα εδάφη που καλλιεργούμε. Και δεν θα μας προστατεύσει κανείς διότι οι επιπτώσεις των προϊόντων αυτών δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η γεωργία. Πρέπει να περάσουμε σε μια διαδικασία που θα επιτρέπει να μην βλάπτουμε ούτε τους καταναλωτές, ούτε το περιβάλλον, ούτε το... τους γεωργούς. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, στην έκθεση αυτή για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων γίνεται πολλής λόγος για την ε, ολοκληρωμένη ε, διαχείριση των ε, παρασιτοκτόνων. Ωστόσο, η έκθεση στην ουσία παρεμβαίνει σε κάποιους γεωργούς στην Ένωση ότι πρέπει πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι όταν έχουμε να συζητήσουμε με θέματα επιλογής φυτών πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία βελτίωσης και των επιλογών που δεν είναι εύκολο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία συχνά δεν επιτρέπει την επιλογή ποικιλιών. Ταυτόχρονα, η οδηγία για τα νητρικά της Ένωσης επιτρέπει, παροτρύνει τη χρήση τεχνητών και όχι φυτικών ε, λιπασμάτων λόγω μέτρων ε, βελτίωσης της πράσινης γεωργίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα την ε, μεγάλη ποσότητα φυσικών νητρικών που διαθέτουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσουμε την διαδικασία χορήγηση αδειών στους γεωργού για να μπορούν να αντιμετωπίσουν γρήγορα τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, 1,5 λεπτό. Κάμπ. Πρόεδρε, η βιωσιμότητα και η λέξη βιωσιμότητα, ορθολογική χρήση και η λέξη γεωργικό φάρμακα είναι αντιφατικές Δυστυχώς εξορισμού τα γεωργικά φάρμακα δεν είναι βιώσιμα ορθολογικά. Τα και τα βρίσκουμε στο έδαφος, στο σώμα, ε, παντού στον κόσμο. Τα γεωργικά φάρμακα επιβαρύνουν την βιοπικιλότητα και αυτό έχει αποδειχθεί. Ε, μιλάμε για διαδικασία εξαφάνισης ενός μεγάλου αριθμού εντόνων, εντόμων απειλούνται, απειλείται σοβαρά η βιοπικιλότητα που έχουν η εξαφάνιση των εντόμων οδηγεί σε ε, αλυσιδωτές αντιδράσεις στα πτηνά αλλά και στην τροφή των ανθρώπων. Η μελέτη αυτή λέει ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι μία από τις βασικές αιτίες Τη μείωση τη βιοπικιλότητα. Άρα το θέμα δεν είναι πώ θα χρησιμοποιούμε οθολογικά τα παρασιτοκτόνα, αλλά πώ θα έχουμε μια γεωργία και έναν τρόπο παραγωγή που θα είναι πραγματικά βιώσιμοι, θα προστατεύουν το, περιβάλλον πρέπει υπολείμματα. εμει βρισκόμαστε στο ξεκίνημα επιδοτήσει τη διαδικασια και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργήσει τι επιδοτησει ε, στη γεωργική παραγωγή. Ευχαριστώ Χόρσλινγκ, δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, το όνομα της έκθεσης ε, είναι ήδη ε, απατηλό. Δεν υπάρχει βιώσιμη χρήση των παραστοκτώνων. Πρέπει να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Να έχουμε μια στρατηγική για τη στρατηγική κατάργησή τους. Και είπατε, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω σχεδίων για την μείωση της χρήσης. Και δεν επετεύχθη τίποτα. Μόνο δύο κράτη-μέλη λέτε ότι έχουν τέτοια σχέδια για τη μείωση. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη αντί για αυτό. Το ανέφερε ο συνάδελφος χρησιμοποιούνται νέο, νέο νοικοτινοειδή, παρά το ότι απαγορεύονται. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Αυτό είναι το έσχος. Πώς είναι δυνατόν να αγνοούν τα κράτη-μέλη την απαγόρευση. Έχουμε τη συζήτηση πάντα για την κλειφωσάτη και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Για τις επιπτώσεις που έχει. Βεβαίως πρέπει να μειωθεί η χρήση της. Λέμε, αλλά παρόλα αυτά αυξάνεται σε ορισμένα κράτη-μέλη. Παρά το ότι υπάρχουν αλλακτικές λύσεις. Η βιολογική γεωργία αποδεικνύει ότι μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτές τις ουσίες. Πρέπει να επανέλθουμε σε μηχανικές μεθόδους. Πρέπει να έχουμε ε, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε αυτό. Αλλά βεβαίως υπάρχουν τεράστια συμφέροντα. Υπάρχει η βιομηχανία που θέλει να βγάλει παραδάκι πουλώντας αυτά τα προϊόντα. Χθες ε, δημοσιεύτηκε μια μελέτη που αποδεικνύει πόσο μειούνται τα είδη. Δεν μας έχει μείνει χρόνος. Πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Και δεν αρκεί να πούμε ότι κάπου και σε κάποιες περιπτώσεις θα μειώσουμε ε, λίγο τη χρήση. Πρέπει να παγορευτούν. Η μελέτη λέει ότι ε, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν το 70% των εντόμων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει και δεν το κάνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε για λεπτομέρειες, για μικροπράγματα, για ακριβή γεωργία, precision farming. Αυτά δεν επαρκούν. Αυτό είναι λίγο καλύτερη τεχνική. Πρέπει να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε πλήρως τη χρήση των ε, ε, προϊόντων αυτών ε, υπέρ και του περιβάλλοντος και των καταναλωτών και των γεωργών. Ντορνανό. Ένα λεπτό για το EFDD. Η κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στη ε, Γαλλία πολλοί έχουν ε, υποστεί τροφική δηλητηρίαση από τα παρασιτοκτόνα. Δυστυχώς πολλοί κλείνουν τα μάτια μπροστά σε αυτό τον ε, υγειονομικό κίνδυνο χωρίς προηγούμενα. Ακόμα και ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε για προϊόντα τα οποία δεν είναι καρκινογόνα, κάτι το οποίο σοκάρισε την κοινή γνώμη. Υπάρχει, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ε, που σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα. Το άρθρο 31 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη βάση αυτού και στην περίπτωση των γεωργών, εάν υπάρχουν συνέπειες, αυτό αφορά το ρυθμό παραγωγικότητας που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι γίγαντες ε, της βιομηχανίας τροφίμων ε, κερδίζουν ε, εκατομμύρια. Νομίζω ότι έτσι δεν επιλύεται το ζήτημα. Μόνο αν βγούμε από αυτό επιλύεται. Ο κύριος Σκοτά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν και συμμερίζομαι την, ε, τα συμπεράσματα της εισηγήτριας για τη μείωση των παρασιτοκτόνων, έτσι ώστε να βελτιωθούν και τα εθνικά προγράμματα δράσης, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της Οδηγίας 128-2009 και του νέου μοντέλου που αφορά την ΚΑΠ. Εάν μιλήσουμε Εάν λάβουμε υπόψη τους στόχους μείωσης των φυτοφαρμάκων, αυτό δεν βοηθάει την εφαρμογή της ΚΑΠ. Θα μπορούσε να πλήξει την αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης ε, δυνάμει της οδηγίας 128 κάθετος 2009. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο χαλαρό σύστημα εφαρμογής της ΚΑΠ, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να φτάσουν σε στρατηγικές παρέμβασεις και όχι σε στενή διαχείριση της ΚΑΠ. Έτσι θα ήταν πιο αποδοτικά και τα εθνικά προγράμματα δράσης. Ακούσαμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Οι υπόλοιποι αγωγητές τώρα. Λίντς, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει να υπάρχει μια ε, αξιόπιστη δυνατότητα έγκρισης και χρήσης των ε, παρεστοκτόνων. Ακούσαμε την έκθεση στις αρχές του χρόνου για την ειδική διαδικασία έγκρισης. Τώρα κάνουμε άλλο ένα βήμα για την βιώσιμη χρήση των προϊόντων αυτών. Εγώ μεγάλωσα σε κτήμα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα και ξέρω πόσο, σωστή είναι, πόσο σημαντική είναι η σωστή χρήση τους. Θεωρώ ότι η υπεύθυνη χρήση των παραστοκτώνων πρέπει να είναι η σωστή προσέγγιση. Βεβαίω πρέπει να υπάρξει και καινοτομία, να βρούμε νέες ουσίες που να είναι πιο αποτελεσματικές και λιγότερο επιβλαβείς. Το δεύτερο είναι η κατάρτιση. Η γεωργία, οι γεωργοί μας δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Παράλληλα, θα πρέπει να μειωθεί η ιδιωτική χρήση. Δεν καταλαβαίνω Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί για παράδειγμα κάποιος τόσο πολλά προϊόντα για το γρασίδι του ενώ απαγορεύεται στο γεωργό η χρήση. Θεωρώ λοιπόν επίσης ότι η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία θα βοηθήσει τη γεωργία και θα οδηγήσει σε πιο περιορισμένη χρήση. Αυτό που δεν αναφέρει ο Σάλφος Χόσλινγκ είναι ότι και η βιολογική γεωργία έχει προβλήματα. Και έχει πολύ χαμηλότερη απόδοση. Η βιολογική γεωργία δεν μπορεί να διασφαλίσει την επιστηστική ασφάλεια που πρέπει και αυτή να μας ενδιαφέρει και ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντριέ. Έχετε, α, θέλετε μπλε κάρτα. <coughs> Σε Για τον κύριο Λίνς. Υπάρχει μπλε κάρτα. Ένα λεπτό κύριε Αντριέ. Σκοτ Κάτο, ερώτηση παρακαλώ. Πού είναι, πού είναι. Εδώ, εδώ. Κύριε, ο κύριος Λίνς ε, επέκρινε ε, τον ε, κύριο Χόισλινγκ γιατί μίλησε για θιούχο χαλκό, ο οποίος χρησιμοποιείται. Το 58% των πεταλούδων και άλλων υπτάμενων ειδών έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε η επόμενη, ε, το επόμενο είδος ε, υποεξαφάνιση. Απάντηση, κύριε Λίνς. Ευχαριστώ. Μα δεν ήταν ερώτηση. Ήταν περισσότερο σχόλιο. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Τι θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε το βασικό θέμα είναι ε, ότι η ποσότητα κάνει κάτι να είναι δηλητήριο. Είτε μιλάμε για παραστοκτόνα, είτε για εντομοκτόνα, είτε για μικητοκτόνα, είτε για οτιδήποτε. Το βασικό είναι η δόση. Έχω την εντύπωση ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό πάντα όλοι οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριο Σάντριο, ενάμιση. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στις 25 Ιανουαρίου τρέχοντος οι Αρχή κρατών και κυβερνήσεων επιτέλους συμφώνησαν να υπάρχουν ε, δείκτες, εναρμονισμένοι δείκτες ε, κινδύνου. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά παράλληλα, την ίδια ημερομηνία, οι εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών δεν ήταν σε θέση να εγκρίνουν τις καθεντήρες γραμμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλουν να προστατεύσουν τους επικονιαστές από, τα, από τη βλάβη που δημιουργούν τα παραστοκτόνα. Η αλήθεια είναι ότι το 2013 ήδη 25 φορές έχει προτείνει η κράτη-μέλη. Από το 2013 έχει προτείνει πώς να προστατεύουμε καλύτερα τις μέλισσες από τα παραστοκτόνα; Το 40% των ντόμων έχουν εξαφανιστεί την τελευταία δεκαετία και σε ορισμένε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πεθάνει το 80% των μελισσών. Η εντατική γεωργία ευθύνεται για αυτήν την παρακμή και παράλληλα η τρομερή χρήση, η υπερβολική χρήση παραστοκτόνων. Οι αργοί κρατών και κυβερνήσεων κρύβονται πίσω από αποφάσει που υποτίθεται πω είναι ευρωπαϊκέ, ενώ δεν είναι. Ενώ είναι οι δικέ του αποφάσει. Η πρόοδο που έχει σημειωθεί για την βιώσιμη χρήση παραστοκτόνων είναι ανεπαρκή. Τρομερά ανεπαρκή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων. Πρέπει να τελειώσει αυτή η υποκρισία από τα κράτη-μέλη για τα παραστοκτώνα στην ουσία αυτό που κάνει είναι να βοηθάει τις ε, πολυεθνικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χτυπήσει το, τη γροθιά στο τραπέζι, να πετύσει τα κράτη-μέλη, να λογοδοτήσουν και να ε, ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση. Είναι θέμα υγείας των 500 εκατομμυρίων των πολιτών της Ένωσης. Μιούλερ, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να υπάρχει βιώσιμη γεωργία η ολοκληρωμένη προστασία από το παράστα είναι υποχρεωτική και πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Η έκθεση στέλνει το σωστό μήνυμα. Αλλά κάτι με ανησυχεί. Παραγγείλαμε μόνο μία μελέτη και θεωρούμε ότι για την μείωση των ειδών των εντόμων φταίει μόνο η γεωργία. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στο επίπεδο ποιότητας που θα έπρεπε να έχουμε στις εργασίες μας. Το γεγονός είναι ότι σε αυτή τη μελέτη είχαν πάρα πολλούς δείκτες για αυτή τη μελέτη και μόνο πολύ λίγοι ε, στηρίζουν τα αποτελέσματά τους. Είναι πολύ συζητήσιμα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Η Γεωργία είναι μόνο ένα από τα διάφορα αίτια που αναφέρει και αυτή ήδη η μελέτη. Μας ανησυχεί βεβαίως αυτό, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά κυρίως πρέπει να κάνουμε περισσότερη έρευνα. Θεωρώ ότι αυτό, ε, δηλαδή η προστασία των ειδών, είναι καθήκον όλων μας και του καθενός μας. Και θα έπρεπε, για παράδειγμα, αντί να έχουμε πολλά φυτά που θέλουν πολλά τέτοια προϊόντα, να έχουμε περισσότερα, περισσότερες πέτρες στους κήπους μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, η οδηγία του 2009 για την χρήση των παρασιτοκτόνων με συμβατό τρόπο με την βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ υπήρχαν σαφείς συνεκτικοί στόχοι και παρότρινε προς την μείωση των παρασυντοκτώνων και την χρήση εναλλακτικών τρόπων. Ωστόσο, η Κομισιόν καθυστέρησε τρία χρόνια για την αξιολόγηση. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι αποτελεί αποτυχία. Γιατί όταν δείτε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας για το Περιβάλλον, βλέπουμε αύξηση 10 με 20% της ζήτησης παρασιτοκτόνων. Ταυτόχρονα και αντίθετα από αυτά που λένε οι συνάδελφοι, βλέπουμε ότι στην βιοπικιλότητα υπάρχει ε, τελείω, μεγάλη μείωση των ασπόνδυλων, ε, ε του οικοσυστήματος, μείωση του αριθμού των πτηνών. Τι θέλουμε. Θέλουμε την καταστροφή της, της ζωής η Επιτροπή και θέλω και το λέει η έκθεση η Επιτροπή πρέπει να παροτρύνει, να ενθαρρύνει τη χρήση των εναλλακτικών με χρηματοδότηση, ενίσχυση της βιώσιμης ε, γεωργίας. Που σημαίνει χωρίς χημικά προϊόντα, χωρίς παραστοκτών. Αυτό είναι το σημαντικό κύριε Επίτροπε. Όχι το αντίστροφο. Πελιτσίνη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση κατά την απόψή μας είναι καλή διότι πρώτον προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα και το περιβάλλον από τους κινδύνους των παρασυντοκτώνων. Μπορεί να βελτιωθεί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ορθολογική χρήση των παρασυντοκτώνων αν δεν δούμε ολόκληρη την, ολόκληρο κύκλο ζωή ε, των προϊόντων αυτών από τη δημιουργία, τη θέση στην αγορά μέχρι την εξάλληψη των υπολοιμάτων. Αν δείτε τις πρακτικές ε, τον, αν δεν αντιμετωπίσουμε τις πρακτικές των απομιμήσεων ε, τα, των εισαγωγών στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να και αν δεν ε, ενισχύσουμε την ρύθμιση, την νομοθετική ρύθμιση και για τους γεωργούς, ε, επιτρέποντας την, απαγορεύοντας την χρήση προϊόντων που περιλαμβάνουν απαγορευμένες ουσίες. Αυτό δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό στην Ευρώπη και επιβαρύνει την ευρωπαϊκή γεωργία άγνιο. Ένα λεπτό. Είναι πολύ της μόδας η αντίρρηση στα παραστοκτόνα. Ορισμένοι λένε ότι είναι θέμα δημόσιας υγείας. Υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία εδώ και 30 χρόνια ε, χρησιμοποιούν ε, και τη συγκεντρωμένη αυτή η ύλη και επίσης την ψεκάζουν και κάποια προϊόντα που χρησιμοποιούσαν πριν από 20 χρόνια ήταν ε, βεβαίως απογορέθηκαν λόγω τοξικών. Όλοι λοιπόν ε, όσοι τα έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ και 30 χρόνια θα πρέπει να έχουμε πεθάνει αν είναι να πιστέψουμε την κινδυνολογία των πρασίνων. Ε, τώρα όσον αφορά την επίπτωση στο περιβάλλον. Βεβαίως αν τα χρησιμοποιήσουμε εντατικά θα ε, κάνουμε μια και στο περιβάλλον και στα ύδατα. Όμως η χρήση τους βοήθησε να θρέψουμε τον πλανήτη η ε, βιολογική γεωργία δεν το επιτρέπει. Και ο κλάδος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μειώσει τη χρήση μέσω τη ε, δημιουργία νέων ειδών που χρειάζονται λιγότερα παραστοκτόνια. Αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα των πρασίνων σε αυτή την ε, επιτυχή τεχνολογία είναι να τα απαγορεύσει αυτά τα νέα είδη. Δεν είναι δυνατόν να έχετε και την πίτα ολόκληρη τόσο φιλοχορτάτο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντουελάε, 1,5 λεπτό. Συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Στην Ολομέλεια συζητάμε συχνά το θέμα των παραστοκτόνων. Εκ νέου η, η χρησιμοποιείται το παραστοκτόνο για να φοβήσει τον κόσμο. Θέλω να πω ότι από την αρχή της θητείας μου φρόντισα να, να τονίσω ότι οι πρώτοι οικολόγοι είναι οι γεωργοί. Οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν την σοβαρότητα και την ασφάλεια τη χρήση των προϊόντων αυτών. Αυτό πρέπει να είναι η βάση των αποφάσεών μα. Πρέπει η προσέγγιση μα να είναι θετική για τον ρόλο τη βιολογική γεωργίας και την προστασία της γεωργίας του περιβάλλοντος από τη γεωργία. Οι γεωργοί πρέπει να συνοδεύονται στις προσπάθειές τους προστασίας του περιβάλλοντος και να βρούμε λύσεις που θα είναι προσαρμοσμένες σε κάθε κατηγορία γεωργίας. Είτε είναι φυτοφαρμακευτική προϊόντα φυσικά ή συνθετικά ή χρήσης εναλλακτικών μεθόδων. Ο σεβασμός της προσέγγισης αυτής προϋποθέτει και θυμίζω αυτό σε όλους ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι πολιτική γεωργίας κατά βάση, όχι περιβαλλοντική πολιτική. Πρέπει να συνοδεύει τους γεωργούς προς την διπλή επίδοση και γεωργική και περιβαλλοντική η κοινή γεωργική πολιτική θα είναι επιτυχής μόνο αν είναι και βιώσιμη. Αλλιώς δεν θα υπάρξει. Ευχαριστώ. Κάντεμπαχ, κυρία Κάντεμπαχ, ένα λεπτό. Πρόεδρε Επίτροπε, δεν είμαστε κατά των γεωργών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η προστασία των φυτών είναι αναγκαία άμα θέλουμε να παράγουμε προϊόντα. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τα φυτά. Και είναι σαφές ότι δεν είναι η μόνη μέθοδος προστασίας των φυτών η μαζική χρήση παραστοκτόνων. Υπάρχουν αλλακτικές δυνατότητες. Υπάρχουν άλλες φυσιολογικές δυνατότητες. Υπάρχουν λιγότερο επικίνδυνα παραστοκτόνα. Υπάρχουν τόσο πολλές αλλακτικές λύσεις σήμερα και αυτό το αναγνωρίζουν ε, οι επιστήμονες, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το εφαρμόζουν επαρκώς και δεν ελέγχουν και δεν επιβάλλουν κυρώσεις όταν υπάρχει ε, υπερβολική χρήση παραστοκτώνων. Τα κράτη-μέλη κάνουν διάφορες εξαιρέσεις που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση των νέων νοικοτινοειδών που θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Θέλουμε να παράγουμε για την Ευρώπη τρόφιμα που να είναι ασφαλή, να είναι υγιή, που να μην βλάπτουν το περιβάλλον, που δεν θα καταστρέφουν την βιοπικιλότητα. Η έκθεση καταδεικνύει πολλές νέες δυνατότητες. Θέλουμε μια νέα ευρωπαϊκή γεωργία και αυτή πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια νέα κοινή γεωργική πολιτική. Δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά χωριστά. Ευχαριστώ, Σκοτ Κέιτο. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εάν δούμε την επικίνδυνη κατάσταση των εντόμων, γιατί το 40% κινδυνεύει με εξάλληψη, ενώ ε, ο πληθυσμός των εντόμων μειώνεται κατά 2,5% ετησίως, αυτό ε, οφείλεται πολύ στην υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Το έχουν πει και οι επιστήμονες. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τα τοξικώς επικίνδυνα παρασιτοκτόνα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει άμεσα αντί να κάνουμε απλώς υποσχέσεις, θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα πλέον τοξικά φυτοφάρμακα έτσι ώστε να προωθήσουμε την, τις οργανικές καλλιέργειες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το οικοσύστημα, εάν λάβουμε υπόψη τον πληθυσμό εντόμων, τους επικονιαστές και ούτω καθεξής. Διαφορετικά θα υπάρχει δραστική μείωση αυτών των πληθυσμών και θα μείνουμε πίσω. Αγιούσο, Πιλάρ, ένα λεπτό. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους στόχους της οδηγίας του 2009 για τα βιώσιμα φυτοφάρμακα και τη χρήση τους. Τα ε, φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να είναι σίγουρα και να υπάρχουν πολύ λίγα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. Γι' αυτό οι γεωργοί έχουν πολλούς περιορισμούς όταν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και βρίσκονται σε μειονεκτική ε, θέση σε σχέση με φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται από άλλα κράτη-μέλη, μάλλον από τρίτες χώρες. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα νέα παράσιτα των καλλιεργιών και να δούμε τι γίνεται με τα παράσιτα τα οποία προέρχονται από έξω. Καλωσορίζω αυτή την έκθεση, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη βιώσιμη χρήση των ε, παρασιτοκτόνων, διότι έχουν μεγάλη σημασία για τη γεωργία. Ντόρφμαν, Herbert, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Ε, πρέπει να είναι προσεκτικό κανεί να χρησιμοποιεί χημικά προϊόντα. Αυτό για τη γεωργία, αλλά και για την ε, υγεία, την ιατρική. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και την προσεκτική χρήση των φαρμάκων. Δεν πρέπει λοιπόν να κατηγορούμε τον Α ή τον Β. Πολλοί είπαν ότι χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παρασιτών. Θέλουμε να έχουμε καλύτερα ε, φυτοφάρμακα με μικρότερη ε, επικινδυνότητα και νομίζω ότι έχουν γίνει προτάσεις για το πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν έχουν γίνει πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη, ιδίω και από δημόσιου ερευνητικού οργανισμού και καλύτερε τεχνικέ χρήσει και πιο ε, ανθεκτικά φυτά. Κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε όλο και περισσότερα παράσιτα που έρχονται στο, από το εξωτερικό. Έχουμε διάφορα είδη, για παράδειγμα, μυγών που καταστρέφουν τα κεράσια. Ε, νομίζω ότι αν προσέχαμε καλύτερα τα σύνορά μας ε, θα είχαμε αποφύγει και μερικά από αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε τώρα. Να ξεκινήσουμε. Καπούτο. Νικόλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έγκριση από πλευρά Κοινοβουλίου του ψηφίσματο τη ε, Ειδική Επιτροπή ΠΕΣΤ ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ενεργοποίηση μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του κανονισμού για, την, για, τη, για τα φυτογειονομικά προϊόντα που επιτρέπει την χρήση ε, αυλαβών παρασιτοκτόνων, δηλαδή που δεν βλάπτουν ε, ζώα ή το περιβάλλον. Η προστασία ωστόσο πρέπει να συμπληρωθεί με μια σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τα παραστοκτόνα που πρέπει να είναι εργαλείο να βοηθήσουμε τους γεωργούς να μειώσουν την εξάρτηση από τα παραστοκτόνα αντικαθιστώντας την εξάρτηση αυτή με προϊόντα βιώσιμα και συμβατά με την οικολογική γεωργία. Για να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες και δεδομένης της τωρινής προστασίας των κατοίκων στην περιοχή αυτή πρέπει επίσης να είναι ένα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, αυτό έχουν στόχο οι τροπολογίες 24 και 44 που προέκυψαν από μια σύνοδο, από μια συνάντηση που και που ζητούν την απαγόρευση της χρήσης ε, παραστοκτώνων όταν βρισκόμαστε κοντά σε σπίτια, νοσοκομεία, ε, παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. Grazie, νομίζω ότι από τη συζήτηση έχει αναδειχθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την χρήση των φυτοφαρμάκων πρόβλημα βεβαίως που αφορά την υγεία και των ανθρώπων και φυσικά την υγεία των ζώων. εγώ κύριε ανδρουικάητη θα ήθελα να θέσω ένα άλλο θέμα διότι συζητούμε για τη χρήση των φυτοφαρμάκων εντός της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά έχουμε αθρώες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από πλευράς τουρκίας και εκεί πέρα η χρήση των φυτοφαρμάκων είναι ανεξέλεγκτη. έχουμε φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων από την τουρκία που απαγορεύονται και όμως αυτά τα προϊόντα εισάγονται πλέον στην ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. επομένως τι προστασία υπάρχει για τους ίδιους τους καταναλωτές. έχουμε ελληνοποίηση γάλακτος το οποίο εισάγεται από την αλβανία ούτε εκεί έχουμε έλεγχο φυτοϊγειονομικό. έχουμε αθρώα εισαγωγή κρεάτων παράνομα από τα σκόπια ούτε και εκεί έχουμε έλεγχο του τι είδους ε, ουσίες χρησιμοποιούν. άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακούσαμε πάρα πολλά σήμερα για την βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και ιδιαίτερα οι αγρότες με το γεγονός ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε την Οδηγία 128 κάθετος 2009 θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι και τα συνοδευτικά μέτρα, αλλά δυστυχώς τα εθνικά προγράμματα δράσης δεν έχουν μετρήσιμους στόχους. Θα πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να έχουν καλύτερη στοχοθέτηση θα πρέπει να έχουν και περισσότερους πόρους. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας των γεών, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις, επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ, ε, λέει ο κύριος Φεραίρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, ουσιαστικά θέματα με την χρήση των ε, παρασιτοκτόνων. Η ΚΑΠ και οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλουν παραγωγικά μοντέλα που σχετίζονται με τις ε, αμετροπείς εξαγωγές. Άρα οι ίδιες πολιτικές είναι ολέθριες για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που έχουν μεγάλη σημασία για την διατροφική ασφάλεια των κρατών. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος της χρήσης των παρασιτοκτόνων και να χρησιμοποιήσουμε μέσα χαμηλότερου κινδύνου, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε τα παραγωγικά μοντέλα και τις συναφείς πολιτικές. Ο κύριος Βιτίδιος. Ε, ο ρόλος των φυτοφαρμάκων για την ε, παραγωγή της Ευρώπης είναι σημαντικός, διότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ε, κινδύνων που προσβάλλουν τα φυτά και συντελούν στην υγεία των φυτών. Όμως μερικά από αυτά εισέρχονται στον υδροφόρο ορίζοντα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στα οικοσυστήματα. Επιπλέον, όταν παραμένουν κατάλοιπα φυτοπαρμάκων επάνω σε τρόφιμα, τίθεται σε κίνδυνο ε, η υγεία των ανθρώπων όσων κατοικούν σε γεωργικές περιοχές, ε, των καταναλωτών αλλά και ακόμη και των περαστικών καθώς επίσης και τα υπολείμματα στις ζωοτροφές αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων. Υπάρχει μια υπόνοια ότι ε, ορισμένα φυτοφάρμακα ευθύνονται για ενδοκρινολογικές διαταραχές. Όλα αυτά επιβάλλουν την υποχρέωση τόσο στα έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν και να κατάλληλουν προσπάθειες για να χρησιμοποιείται με ορθολογιστικό τρόπο τα φυτοφάρμακα. Ε, πρέπει να περιοριστεί η χρήση των φυτοφαρμάκων και να επιλεγούν ε, όχι χημικές αλλά βιολογικές μέθοδοι. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τα φυτοφάρμακα, να προστατεύσει τους καταναλωτές από φυτοφάρμακα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες. Φαρία. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει σωστή η διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως ε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει ε, δύο ποικιλομορφία αλλά επίσης ολέθρια παρασίτοκτόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θρέψει κανείς επτά δις στον κόσμο αυτό και πολλές φορές ε, γίνεται χρήση παρασίτοκτόνων που είναι εύκολα στη χρήση χωρίς να, να αποτιμηθούν οι κίνδυνοι. Πρόκειται για 500 τέτοιες ε, δραστικές ουσίες οι οποίες ε, δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε βιώσιμες εναλλακτικές για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και οι αγρότες τις ε, πιο αποδοτικές λύσεις βραχυχρόνια. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Βεβαίως ε, σήμερα μιλάμε για ένα ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει να είμαστε και ορθολογικοί. Όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει όμως να δούμε ποια είναι και τα ενδεχόμενα σενάρια. Δεν μπορούμε να αποδεκατήσουμε τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει και μία τελωνιακή αρχή η οποία να ελέγχει όλα τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κομμάτι-κομμάτι. Θα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν αυτό το πλαίσιο, αλλά Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να εναρμονίσουμε αυτά τα μέσα και να υπάρχει και εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα θα πρέπει να επαληθεύονται σε σχέση με την τοξικότητά τους. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε επενδύσεις στην ε, έρευνα και στην καινοτομία. Ε, κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Θέλω να διευκρινίσω ποια είναι η προσέγγιση μου. Στηρίζω την προστασία της υγείας ε, των πολιτών μας. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τους παραγωγούς, τους γεωργούς μας, για τους οποίους ε, είναι αναγκαία τα φυτοφάρμακα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια πίεση για την μείωση της χρήσης τους και για την απαγόρευση ορισμένων, ιδίως αυτών που είναι καρκινογενή. Αυτό βεβαίως έχει έννοια. Αυτό το κατέδειξε και μία έκθεση της ΕΦΣΑ που δείχνει ότι ε, πολλά ε, φυτοφάρμακα δεν αφήνουν ε, τελικά ίχνη. Βεβαίως πρέπει να απαγορεύσουμε το πιο επικίνδυνα, αλλά να στραφούμε προς τα λιγότερο επικίνδυνα και κυρίως βεβαίως να αντιμετωπίσουμε και τις αγωγές επικίνδυνων τέτοιων φαρμάκων. Ζωάννα. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να γίνει ε, λελογισμένη χρήση των ε, παρασιτοκτόνων για να μειώσουμε βεβαίως ε, και τις ασθένειες, αλλά να μην μπουν αυτά τα προϊόντα στον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι ώστε να πλήξουν και άλλους πληθυσμούς καθώς και τους ε, υδάτινους σπόρους. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις ως προς τα νεονικοτινοειδή. Θα πρέπει να απαγορευτεί πλήρως η χρήση τους. Ό,τι ισχύει στη ε, Γερμανία θα πρέπει να ισχύει και στη Βουλγαρία. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε παρασιτοκτόνα, τα οποία όμως να μην έχουν επικίνδυνες δραστικές ουσίες, έτσι ώστε να μην πλήξουμε ούτε τον άνθρωπο, ούτε το περιβάλλον. Να υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες στο μέτρο του δυνατού. Ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, λέμε πολλά για την ε, χρήση φυτοφαρμάκων. Είχαμε και μια ειδική έκθεση, μια ειδική επιτροπή μάλιστα. Σήμερα έχουμε και αυτήν την ε, έκθεση. Ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερα φυτοφάρμακα και κυρίως ε, να απαγορεύσουμε τα πιο επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Γι' αυτό Πρέπει να προτιμήσουμε την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ε, παρασίτων, νέες τεχνικές για τον ψεκασμό να ε, προωθήσουμε και να βοηθήσουμε και όσους είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν πρώτοι αυτές τις μεθόδους. Κοιτάξτε, για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη θα συνεχιστεί στη γεωργία η χρήση των ε, παρασιτοκτόνων. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την ακριβή γεωργία. Δηλαδή, συγκεκριμένες τεχνικές που μας επιτρέπουν να καταστρέφουμε τα παράσιτα ε, με άλλες μεθόδους. Να τα καταστρέφουμε με πιο ε, οικολογικές μεθόδους. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye, οπότε να επανέλθουμε προς τον Επίτροπο κύριο Άντριου Κάιτης για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα πολύ προσεκτικά και άκουσα πολλά λογικά επιχειρήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υπάρχει βιώσιμη χρήση των παραστακτώνων και η βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας. Αλλά να αντιδράσω σε κάποια τα οποία υπόθηκαν. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Φλόρεντς όταν μιλάει για την κατάρτιση. Τώρα υπάρχουν πολλές νέες ε, γεωργικές τεχνικές. Πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να προσέξουν περισσότερο την κατάρτιση. Εφόσον τώρα οι γεωργοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνικές για τη χρήση των ε, φυτοφαρμάκων και για τις εξαιρέσεις. εξαιρέσεις πρέπει να είναι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας. Η Επιτροπή Βεβαίως ε, τα εξετάζει όλα αυτά πολύ επισταμένος και έχουμε εισαγάγει αυστηρά μέτρα όπου απαιτούμε τα κράτη-μέλη να αιτιολογούν τις εξαιρέσεις να δούμε πώς μπορούν να μειωθούν, να καταργηθούν και έχουμε ένα συνεχή διάλογο με ορισμένα κράτη-μέλη για αυτές τις εξαιρέσεις, οι οποίες όμως επιτρέπονται από τον νόμο. Πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο όμως με αυτές. Ορισμένοι Είπατε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση ε, λιγότερο επικινδύνων φυτοφαρμάκων. Έχουμε πολλούς νέους κανόνες, πολλές βελτιώσεις διαδικασίες, ε, ούτως ώστε να υπάρξει ταχεία έγκριση πιο ακινδύνων φυτοφαρμάκων. Υπόθηκε επίσης ότι η βιολογική γεωργία δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες. Όχι. Και στη βιολογική γεωργία κάποια χημικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα ο ε, ε, χαλκός. Ο θηκός χαλκός ε, ε, είναι καρκινογενής, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να μην ε, εξαπατούμε τους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι όλα τα είδη γεωργίας χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και όλες οι μέθοδοι χρησιμοποιούν χημικά. Μην δημιουργείτε τεχνητές αντιπαραθέσεις μεταξύ συμβατικής και βιολογικής γεωργίας. Να πείτε την αλήθεια στους καταναλωτές. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, εμείς που ε, καταρτίζουμε τους κανόνες. Ξέρουμε πώς τα διαφορετικά είδη γεωργίας χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία. Και σωστά είπατε ότι ε, δεν είναι εύκολο να υπάρξει η ειδική πλειοψηφία στην μόνιμη Επιτροπή Γεωργίας γιατί τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Και άρα πρέπει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν την πρώτη ανάγνωση για την επιτροπολογία, για τους κανόνες επιτροπολογίας, όπου προτείναμε να υπάρξει διαφάνεια στην διαχείριση των κινδύνων, αλλάζοντας τους κανόνες της ε, επιτροπολογίας, για να είναι τα στοιχεία προσβάσιμα από το κοινό. αλλά εδώ και δύο χρόνια δεν έχει προχωρήσει η πρώτη ανάγνωση. Σας ε, καλώ να το τονίσετε το θέμα αυτό έναντι της κοινή γνώμη. Χαίρομαι που χθε ολοκληρώθηκε ο τριμερής διάλογος για το Γενικό Νόμο για τα Τρόφιμα και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιούσο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην αξιολόγηση των παραστοκτώνων και αυτό είναι ένα μεγάλο επιτεύγμα. Και επίσης ε, ε, προτείνω ε, ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία των φυτών. Κάνουμε πολλές προσπάθειες και δεν υπάρχει βέβαια κανένα τέλειο σύστημα. Η κυρία Ντογνανό είπε ότι αυτοκτονούν πολλοί οι γεωργοί στη Γαλλία. Συναντήθηκα στη Γαλλία με τις γαλλικές αρχές για το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να δουν τι γίνεται πολύ προσεκτικά για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Κάποιοι λένε ότι τα φυτοφάρμακα είναι δηλητήριο. Ναι, τα φάρμακα γενικά, όλα τα φάρμακα είναι δηλητήρια. Αλλά προσέξτε, μην ε, ε υπερβάλλετε. Η Επιτροπή περιμένει την έγκριση του κανονισμού για την χρήση των φυτοφαρμάκων και τα μέγιστα επίπεδα χρήσης. Επίση, θέλουμε να κάνουμε και την αξιολόγηση τη εφαρμογή αυτή τη οδηγίας το 2020 για να δούμε αν είναι επαρκή αυτή η οδηγία. Καλό τα κράτη-μέλη να θέσουν φιλόδοξου στόχου. Υπάρχει σαφέ χρονοδιάγραμμα. Μάλλον πρέπει να θέσουν ένα σαφέ χρονοδιάγραμμα στα εθνικά σχέδια δράση. Πρέπει να αποδείξουν έναν των πολιτών τη δέσμευσή του για τη μείωση των φυτοφαρμάκων λόγω των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σα ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη στήριξή σα για το σημαντικό αυτό θέμα. Προσβλέπω στην έγκριση αυτή τη σημαντική έκθεση από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Γκιούτε Χιούτελαν και του Σκιώδη για τη θαυμάσια ε, συνεργασία και για την πολύ αναλυτική έκθεση. Θα λάβουμε υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης και θα συνεχίσουμε στην πορεία προς μια πιο βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη για να προστατεύσουμε τους ε, συμπολίτες μας, το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τη βιώσιμη γεωργία και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να κλείσει κύριε Ντάλη. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Προφανώς είναι αμφιλεγόμενο θέμα. Η χρήση των παραστικτοκτώνων παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη γιατί βοηθά να διατηρούμε τα φυτά υγιή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και οδηγεί επιτρέπει την μείωση της καταστροφής των φυτών από ζυζάνια και ασθένειες. Ωστόσο, η χρήση των παραστοκτώνων δεν είναι βιώσιμη και όταν δεν είναι βιώσιμη οδηγεί σε απώλεια της βιοπικιλότητας και σε μόλυνση του νερού, επιφανειακού και υπόγειου και του εδάφους. Για τους λόγους αυτούς ανησυχούμε από το ότι από το γεγονός ότι τα ζυζανιοκτώνα μπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου μέσω της αλυσίδας διατροφής. Αυτός είναι ο λόγος που εκφράζονται ανησυχίες ιδίως όταν μιλάμε για περιπτώσεις ατόμων που εκτίθενται σε παρασιτοκτόνα που να έχουν ε, ιδιότητες ε, ενδοκρινοπαρενοχλητικές. Επιπλέον, η χρήση των παρασιτοκτόνων δεν είναι βιώσιμη, δεν είναι συμβατή με τη βιώσιμη γεωργία και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την βιώσιμη γεωργία, την πρόληψη, την χρήση μη χημικών ουσιών, βιολογικούς ελέγχους και προγράμματα χαμηλού κινδύνου. Η έκθεση που συζητούμε τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι δίνει ένα μήνυμα προόδου που μπορώ να συνοψίσω ως εξής. Πρώτον, τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν καλύτερα τα εθνικά σχέδια δράσης προωθώντας μη χημικές εναλλακτικές λύσεις και προϊόντα που προστατεύουν τα φυτά με χαμηλό κίνδυνο. Τα παραστητοκτόνα θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, πάρκα ή κοντά σε έγκυες γυναίκες. Τρίτον, η συλλογή δεδομένων για τα παρασυντοκτόνα και τα υπολείμματά τους θα πρέπει να βελτιωθεί με καλύτερα μέτρα για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας. Θα δίνουμε λοιπόν όλες τις πολιτικές ομάδες να περάσουν ένα ισχυρό μήνυμα προς την κατεύθυνση αυτή στη σημερινή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα. Ολοκληρώνεται η σχετική συζήτηση. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη έκθεση, την έκθεση του κύριου Μπέλετ, για την εφαρμογή της οδηγίας για την διασυνοριακή ετοφαρμακευτική περίθαλψη. Μόλις τελειώσετε να παίρνετε φωτογραφίες κύριε Μπέλετ θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, Καλημερίσω όλους, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Εάν υπάρχει ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε προστιθέμενη αξία, ε, είναι ο τομέας υγείας, ιδιαίτερα στις όμορες περιοχές. Είναι πολύ πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό να πάει κανείς στο νοσοκομείο που είναι στην άλλη πλευρά των συνόρων. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις σπάνιες ασθένειες ή τις χρόνιες ασθένειες που, όπου οι ασθενείς βρίσκουν καλύτερη περίθαλψη στην άλλη πλευρά των συνόρων. Και δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, πολλές φορές ε, γραφειοκρατία, φοβερή γραφειοκρατία, όταν πρέπει να μεταβεί κανείς στο εξωτερικό και δεν ξέρει πότε θα του επιστραφούν τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτά τα προσκόμματα. Η οδηγία για την διασυνοριακή περίθαλψη συντάχθηκε αρχικά το 2011 Υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Πρόκειται για μία έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και υπάρχουν πολλές ε, πρακτικού είδους ε, συστάσεις. Η πρώτη ανάγκη είναι οι πληροφορίες ε, για τους ασθενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, ούτε ξέρουν από που μπορούν να αντλήσουν αυτή την ε, πληροφόρηση. Γι' αυτό ζητήσαμε ενιαίες θηρίδες πληροφόρησης όπου οι ασθενείς μπορούν να λάβουν όλες ε, τις πληροφορίες για την περίθαλψη, επιστροφή ιατρικών εξόδων και ούτω καθεξής. Οι ασθενείς λοιπόν θα πρέπει να έχουν μία σαφή εικόνα για την διασυνοριακή περίθαλψη, διότι αντιμετωπίζουν φοβερή γραφειοκρατία. Νομίζω ότι εδώ μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποτιμά την κατάσταση σε αιτήσια βάση με τη συνδρομή των εθνικών αρχών. Τώρα, σε σχέση με τους ασθενείς, με χρόνιες ασθένειες ή σπάνιες ασθένειες, πολλές φορές χρειάζεται εξειδικευμένη ε, ε, περίθαλψη σε ένα άλλο κράτος μέλος. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε συναφείς πληροφορίες και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνδράμουν με ε, εξειδικευμένα Ινστιτούτα όπου ε, υπάρχει τεχνογνωσία εχμής. Τέλος, ως προς τη ψηφιοποίηση, στον τομέα της ε, υγείας και της ιατρικής περίθαλψης, η ψηφιοποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο βελτίωσης παροχών υπηρεσιών. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσατε για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ελπίζω να το προωθήσετε σύντομα μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Χρειαζόμαστε μία εύρωστη πολιτική και τα, οι πολίτες μας αξίζουν της ε, καλύτερης ε, ιατροφαρμακευτικής ε, περί, περίθαλψης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την υγεία τους. Η κυρία Γκραπίνη από πλευράς ΙΜΚΟ και εγώ υποστηρίζω αυτή την έκθεση, θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς εφαρμόζεται στα κράτη